Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, mes Αγαπητοί συνάδελφοι, Γάλλοι φίλοι, Λοιπόν, μετά την κοινή συνεδρίαση της, ε, με την Επιτροπή Λίβε, τώρα είμαστε πάλι εμείς και εμείς, η Επιτροπή Οικονομικών, και ξεκινάω πρώτα απ' όλα με μια διαβούλευση, εκ νέου διαβούλευση, μια επιστολή έστειλε το Συμβούλιο 21 Ιανουαρίου και μας ενημέρωσε πως η Κορεπέρα επέτυχε πολιτική συμφωνία για τον κανονισμό για τα τέλη και χρεώσεις σε συναλλαγές με κάρτες, το λεγομενο ΜΥΦΔΙΟ. MIF2, και η πρώτη ανάγνωση είχε γίνει στην προηγούμενη θητεία τον Απρίλιο πέρσι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το ενοποιημένο κείμενο της Συμφωνίας ε, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και το είχατε στη διάθεσή σας και τώρα πρέπει να το ψηφίσουμε. αν συμφωνούμε δηλαδή με αυτή την συμφωνία. Πριν το ψηφίσουμε όμως θα δώσω τον λόγο στον εισηγητή μας, ο κύριος Μπι Δεγκαΐν. Πάμπλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Να ζητήσω απλώς την υποστήριξή σας για αυτή την πολύ σημαντική έκθεση μέσω της οποίας θα καταφέρουμε να πληρώνονται λιγότερες προμήθειες ε, από τους ε, Ευρωπαίους φορολογουμένους όταν κάνουν ε, συναλλαγές με πιστοτικές κάρτες. Να ευχαριστήσω τους κοιόδης συγητές και τους συντονιστές και φυσικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πριν περάσουμε στην ψηφοφορία να ρωτήσω εάν έχετε όλοι τις κάρτες σας εδώ της ψηφοφορίας από ό,τι φαίνεται ναι. Λοιπόν, να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία, να δούμε αν θα παραμείνουν όλοι εντός των ορίων, όλες οι ομάδες. Έξι, πέντε δεν ψήφισαν ακόμα, αναβαίνει ακόμα ο αριθμός των καρτών. Τέσσερι συνάδελφοι έχουν βάλει την κάρτα και δεν ψήφισαν ακόμα. Τώρα είναι όλα καλά. Μάλιστα και λείπει μία συνάδελφος. Κλείνουμε λοιπόν. Όλες οι ομάδες εκπροσωπούνται σωστά. Ονομαστική ψηφοφορία για το αποτέλεσμα λοιπόν της διαπραγμάτευσης για το ΜΥΦ2. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Ναι, ευρεία πλειοψηφία. Στον εισηγητή, ε, συγχαίρω τον εισηγητή και ολόκληρη την διαπραγματευτική ομάδα. Το κείμενο θα πάει τον Απρίλιο στην Ολομέλεια όταν περάσει και από τους γλωσσομαθείς γνωμικούς ε, για να ψηφιστεί. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία για την έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού. Εισηγητής ο κύριος Μέσσερ Σμιτ. Έχετε να πείτε κάτι ή ξεκινάμε απευθείας. Θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ όλους τους κοιόδης εισηγητές ε, που συνέβαλαν σε ένα πνεύμα συμβιβασμού και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να στείλουμε ένα σαφές αν όχι ομόφωνο μήνυμα προς την Κομισιόν για την πολιτική του ανταγωνισμού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ κύριε Μέστερ Σμιτ. Ψηφίζουμε. Συμβαστική Α υπέρ. Κατά. Οχές. Εγκρίνεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές ναι, ας το μια φορά όμως. 64. Αρχίζει η ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Απερίφθη. Συμβαστική Β υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 72. Να επαληθεύσουμε. Επαληθεύουμε την 70 παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. 26-26 απερίφθη λοιπόν. Μα είχα δίκιο. Κυρία συνάδελφε, να με ακολουθείτε άλλη φορά. Μη λέτε μόνο α και αου. Να λέτε αυτό ο γερακή σιωμάτι, ο πρόεδρος. 72 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Να επαληθεύσουμε λοιπόν. 72. Επαλήθευση ηλεκτρονική. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Και εδώ είχε δίκιο ο πρόεδρος. Εγκρίνατε. 73. Έχει καλυφθεί από την συμβαστική ε. 74 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε λοιπόν. 74 αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Συμβαστική C γάμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική D δέλτα. Υπέρ. Κατά. αποχές 84 ε, παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε 85 Πέρας της σοφορίας εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές Έχει απορριφθεί νομίζω, αλλά σε παληθεύσουμε αν δεν έχετε αντίρρηση. 91 αρχίζει η ψηφοφορία. Ε, έχουμε έναν υπεράριθμο από τους σοσιαλιστές δημοκράτες ένας υπεράριθμος από τους σοσιαλιστέ δημοκράτες. Θα πρέπει κάποιο να αποσύρει την κάρτα του. Εντάξει. Πέρα της ψηφοφορία. εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά Αποχέ. απερίφθη Συμβαστική σίγμα F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται, αλλά σε επαληθεύσουμε. F. Σίγμα F. Επαληθεύεται. Αρχής προφορία. πέρας Εγκρίνεται. Και τώρα προχωρώ. 101, 108, συγγνώμη, 108 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 109 υπέρ, κατά, αποχές. Να επαληθεύσουμε 109. Πέρασε. Εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δυστυχώς απερίφθη. Συμβαστική G, Z, υπέρ. Α, σε τμήματα έχουμε εδώ. Λοιπόν, πρώτο τμήμα και μετά δεύτερο. Ψηφίσουμε το πρώτο, παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές. Θα το επαλήθευα. Δεύτερο τμήμα συμβαστικής Z. G. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρασε ψηφοφορίας, απερίφθη. Συνεχίζω λοιπόν στην 119. 119. Συμφωνεί και ο εισηγητής. Στην 119 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ηττα. H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 κατά αποχές εγώ λέω ότι είχε απορριφθεί, αλλά στο επαληθεύσουμε καλύτερα. 126. Επαληθεύουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 127. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 133 υπέρ κατά οι σοσιαλιστές και είναι κατά έτσι άποχες Ας επαληθεύσουμε 133 αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε. 134. Αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά. Άποχες. Με την ίδια πλειοψηφία. 136 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Άρα πάμε στο αρχικό κείμενο της παραγράφου 10 παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική I, λατινικό, θήτα στα ελληνικά, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική J, J στα ελληνικά, υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 153 παρακαλώ, υπέρ, υπέρ. Δεν <laughs> σηκώνω τα άλλα χέρια, κατά. Άποχες, απερίφθη. 154 υπέρ, κατά, άποχες Εγκρίνεται 155 υπέρ κατά άποχες απερίφθη. 156 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά ας ε, επαληθεύσουμε παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Σωστά το είδα. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 158. Εντάξει. 157. έχουμε την 157. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 158. 158. Κατά. Απόχες. Να επαληθεύσουμε και αυτό. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 160 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 161 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 162 υπέρ κατά άποχες απεριφθεί 163 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνατε 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική K για τα α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική L λατινικό για τα β στα ελληνικά υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 168 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 170 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 171 υπέρ κατά αποχές απερίφθη επαληθεύουμε την 171 αυτό θέλετε αρχίζει ψηφοφορία 171 ψήφισαν όλοι πέρας απορρίπτεται 173 υπέρ κατά αποχές να την ξαναδούμε και αυτήν. Τεμπελιάζεται λίγο. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Όχι, όχι η πρώτη σειρά. Λοιπόν, ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. «174. Υπέρ». «Κατά». «Αποχές». Οι πράσινοι δεν έχουν άποψη. Α, δεν σηκώνεται χεράκι. Λοιπόν, δεκτή. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. Νομίζω πως απορρίφθηκε. 176. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. Να την ξαναδούμε. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι γίνεται δεκτή. Δεκτή. Δεκτή. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές Δεκτή. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο λοιπόν της παραγράφου υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να την επαληθεύσουμε την 191 άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας δεκτή 192 υπέρ κατά αποχές δεκτή 193 υπέρ κατά αποχές δεκτή 194 υπέρ κατά αποχές δεκτή 195 υπέρ κατά αποχές δεκτή 196 υπέρ κατά άποχες δεκτή 197 υπέρ κατά άποχες να την επαληθέσουμε άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας δεκτή 198 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 200 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο της παραγράφου 15 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο της παραγράφου 15 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική ε, μη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 206 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί στους φιλελεύθερους. Λοιπόν, επαληθεύουμε την 207. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. 208 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 209 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική νη, νίκος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 211. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. 211 άρχεται η ψηφοφορία. 211. Ό,τι και αν είναι αυτό. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Σαφές. Απορρίπτεται. 212 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 213 υπέρ. Κατά. Συγγνώμη. Έχετε δίκιο. 214 υπέρ 2.14 ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.15 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι γίνεται δεκτή αλλά να τη δούμε 2.15 ψηφίζουμε Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. 216 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 217 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.18 καλύπτεται νομίζω από την F. Πρέπει να ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο. Ηρεμία, ηρεμία, ηρεμία. Θα φτάσουμε. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 18 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Είδες. Λοιπόν, 2.19 υπέρ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μικρός και άπειρος. Κατά, αποχές, να την επαληθεύσουμε. Την 2.19 άρχεται η ψηφοφορία. Α, τώρα είναι πάλι σαφές. Λοιπόν, δεκτή. 2.20. Ναι, ξαφνικά οι δύο μεγάλες ομάδες. Ναι, ναι, εσείς οπωσδήποτε, ναι. Η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα. Λοιπόν. 2.20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να την επαληθεύσουμε. Την 2.20. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική όμικρον. Όλγα. Χωριστή ψηφοφορία. Μέρος πρώτο. Ποιο είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2.25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μπορούμε να την επαληθεύσουμε την 2.25, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται σαφώς. 2.26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2.27. Υπέρ. Κατά. Αποχές Ναι. Καλύπτεται από την 226. Περνάμε λοιπόν στην 230. 2.30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2.31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 232 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή 233 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική π Παύλος υπέρ κατά αποχές Απο... δεκτή 2.39 ε, υπέρ κατά αποχές θα ήθελα να την ξαναδούμε άρχεται η ψηφορία για την 2.39 Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Δεκτή. 2.40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2.41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2.42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική Q λατινικό. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2.47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2.48 υπέρ κατά αποχές με μεγάλη διαφορά δεκτή 2.49 υπέρ κατά με ακόμη μεγαλύτερη διαφορά δεκτή 2.50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.52 υπέρ κατά αποχές Απορρίφτεται. συμβαστική ρο όπως Ριχάρδος υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.56 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική σίγμα Σαμουήλ υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.59 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε την 2.59 άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας δεκτή συμβαστική όπως τάσος υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.62 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 264 υπέρ κατά άποχες θέλω να την ξαναδούμε ε, οι φιλελεύθεροι παρακαλώ να ψηφίζετε λοιπόν άρχεται η σωφορία. εννοώ με το χέρι ε, γιατί δεν σας βλέπω ψήφισαν όλοι πέρας δεκτή Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. 2.65. Υπέρ. Κατά. Μάλιστα. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. 2.65. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίφτεται. 266 υπέρ κατά αποχές δεκτή 267 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο της παραγράφου 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή 273 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό της παραγράφου 27 υπέρ να την επαληθεύσουμε την 273 μάλιστα άρχεται η ψηφοφορία 273 ψήφισαν όλοι πέρας απορρίπτεται και τώρα το αρχικό κείμενο στην 27 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. 274 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 275 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΒΙΧ λατινικό υπέρ κατά Άποχες, εγκρίνεται. 283 υπέρ. Α, μπορούμε να ψηφίσουμε on block. Όχι, εγώ δεν έχω το, την διαπληροφορία στην πληροφορία μου. Πάμε λοιπόν 283 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 284 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 285 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 286 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 287 υπέρ ε μα ήταν σαφές το αποτέλεσμα τι 286 σαφέστατο ό,τι στοίχημα θέλετε κύριε Γκίγκολτ 286 κατόπιν ειδικού αιτήματος των πρασίνων αρχίζουμε την ψηφοφορία 2, 8, 6 286 πέρας τη ψηφοφορίας ότι έκπληξη εγκρίνεται Αυτό είναι το πλεονέκτημα έχει όποιος κάθεται στο Προεδρείο. Βλέπει καλύτερα. Λοιπόν, 287 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στους κανονικούς μας ρυθμούς. Συμβιβαστική τροπολογία W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 τώρα παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 29 επαληθεύουμε. Επαληθεύουμε την 28. Αρχίζει η ψηφοφορία. 28 για όσους δεν καταλαβαίνουν. <coughs> Βαβαρέζικα μου. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. 29 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά αποχές με την αυτή πλειοψηφία εγκρίνεται ε, υπέρ ήταν οι δύο φιλελεύθεροι επαληθεύουμε πάντως 29 υπέρ ψηφίσατε όλοι πέρα της απερίφθη λοιπόν ευχαριστούμε τον κύριο Λάγκεν ε, X, λατινικό, συμβαστική τροπολογία περιθμών. X, υπέρ παρακαλώ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Συμβαστική Y, Y, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές απερίφθη το αρχικό κείμενο στο αιτιολογικό C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ζήτα Z υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές απερίφθη Αλφα, υπέρ Α, ε, ε, κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΑΒ AB υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θεολογικό station 1 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απερίφθη τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απερίφθη το αρχικό κείμενο της ιδεολογικής πρότασης ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παριθμόν ένα υπέρ κατά απόχέ. απεριφθεί Τιολογική πρόταση 3, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τιολογική πρόταση 4, αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θεολογική ε, τροπολογία νομή 4 μια παρατήρηση εκτός μικροφώνου δεν ακούστηκε η 4 λοιπόν τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 5 υπέρ κατά νομίζω ότι αυτό λύθηκε. Αποχές απερίφθη. Έξι, τροπολογία έξι, υπέρ. Ζητώ συγγνώμη, απερίφθη. Πάμε στο πρωτότυπο κείμενο, στο αρχικό κείμενο. Ο κύριο Κολμπέτ δεν ακούγεται χωρί μικρόφωνο, δεν είναι δυνατόν να μεταφραστεί. Χαιρόμαστε πολύ που εδώ, λέει ο πρόεδρο. Η σοφία τη Επιτροπή των Σταματικών Υποθέσεων. Τροπολογία 6, λοιπόν, υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Και έτσι ισχύει ο ίδιος κανόνας φαντάζομαι. Και πάμε στην 7. Υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 8. Υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 9. Υπέρ κατά αποχές απερίφθη 11 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 11 υπέρ κατά αποχές απερίφθη Τεολογική πρόταση 15 αρχικό κείμενο. 16 συγγνώμη αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 14. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. η Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Το αρχικό κείμενο στην 24 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογική σκέψη 25 το αρχικό κείμενο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 18 υπέρ, κατά αποχές. Απερίφθη. Τελογικές προτάσεις 27-41 αρχικό κείμενο υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνονται. Η τροπολογία 19 υπέρ, κατά εποχές. Ας επαληθεύσουμε. Την 19 παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. κρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύω. 20. Αρχίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. 21 παρακαλώ. είπε Κάτσα. Αποχές. έχουμε πάντα βέβαια. Αρχίζουμε την 21, επαληθεύουμε την 21, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα, παράγραφος 10 της Επιτροπής μπορούμε να κάνουμε την ΕΜΚΟ συνολικά. Αμα να μου το λέτε όμως άμα είναι λάθος. Λοιπόν, παράγραφος 1. Υπέρ. Κάτω. Ε, παληθεύουμε. Μάλλον 10 εννοεί ο πρόεδρος. Α, όχι, ε, 1, συγγνώμη. Παράγραφος 1 τη ΣΥΜΚΟ. Αρχής προφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. ΕΜΚΟ παράγραφος 2. Καλά, τώρα ανοίγουμε. Από 2 έως 19 η παράγραφη. Μπορούμε να τα κάνουμε on block. 12. Καλά. Ε, όλες λοιπόν οι υπόλοιπες παράγραφοι πλην τις 12. 2, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19 υπέρ παρακαλώ. Να σηκώσετε τα χέρια σας. Α, κύριε καθηγητά Λούκερν, να, προχα... να προσέχατε. Πρόεδρε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Για το 15, 15 δεν θέλαμε να βάλουμε στην ομπλόξη σου ε, Μα μου είπατε το 12 όμως, τι είναι αυτό. Άντε καλά. Λοιπόν. 2, 7, 8, 9, 10, 12. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 15 τώρα, τη ΣΥΜΚΟ κατά αποχές εγκρίνεται. Τις υπόλοιπες μπορούμε πάλι 18 και 19. Κύριε Σίγητα, σας ευχαριστώ υπέρ της 18-19 λοιπόν. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για να δούμε λοιπόν ονομαστικά το σύνολο της προτάσεως. Ονομαστικά, αρχής ψηφοφορίας. Ψήφισαν οι πάντες. Πέρας. 51 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά, 4 ψήφοι αποχής. Συγχαρητήρια στον ε, εισηγητή μας και στους πολυάριθμους και όδες. Έχουμε να βάλει την ψηφοφορία για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Άρα για τις προφορίες τελειώσαμε προς το παρόν και κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Συνεχίζουμε λοιπόν, παρακαλώ, με την ημερήσια διάταξη. Με τα σημεία 13, 14 και 15 της ημερήσιας διάταξης μαζί αφορούν τις απαλλαγές. Και με χαρά δίνω το λόγο στον εισηγητή. Παρακαλώ όμως ότι μεταξύ Να μην σα ελπίζω να σας ενοχλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, στις κουβεντούλες σας. Ελίζα. Μπριγάδο. Στην απαλλαγή λοιπόν των τριών αρχών. Έχουμε γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Έχω εγώ την τιμή να στάσω τις σχετικές γνωμοδοτήσεις. Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους για τις πολύ άριθμες τροπολογίες 26 για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, 23 για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και 26 για την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Έχουμε να κάνουμε τρεις τομείς που καλύπτω και στις ε, γνωμοδοτήσεις μου. Καταρχάς έχω τον, ε, τους στόχους, τις λειτουργίες, τις προτεραιότητες, την χρηματοδότηση, πρικοδότηση των τριών υπηρεσιών τα ζητήματα των ε, προτύπων χρηματοδότησης. Στο θέμα της Ευρωπαϊκής ε, Αρχής Τραπεζών λαμβάνω υπόψη βέβαια και την έκτακτη έκθεση παριθμών 5 του Ελεκτικού Συνεδρίου για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Εποπτείας στο πλαίσιο της ε, Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης και των δομών των τραπεζικών του Ελεκτικού Συνεδρίου. Έχουμε να κάνουμε βεβαίως με πολλά κοινά ζητήματα που παρατηρούν στα αρχαία πολλές ομάδες. Εκόπτει ο πρόεδρος. Μήπως οι σοσιαλιστές ε, βοηθοί μπορούν να κάνουν τις κουβεντούλες τους πιο ήσυχα ή έξω. Σας καταλαβαίνω, εδώ που βρίσκομαι καταλαβαίνω τι λέτε για να ξέρετε. Έχουμε λοιπόν πολλά σημεία κοινά από τις τροπολογίες που έχουν υποβάλει οι ομάδες. Άρα πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια καλή λύση με τις ψηφοφορίες. έχουμε τον ρόλο των τραπεζών που αναγνωρίζει το σημαντικός, αλλά βέβαια και σαφείς προτεραιότητες που ορίζουμε, ότι λέμε επίσης ότι θα πρέπει να επεκταθεί υπερβολικά η εντολή τους, να διωγγωθεί υπερβολικά. Λέμε ότι χρειάζεται η κατάλληλη ε, οικονομική κάλυψη, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει μια επιταγή εν λευκό, χωρίς καμία εποπτεία στις δραστηριότητες. Να μην ε, διονγκώνονται δηλαδή ο κύκλος των αρμοδιοτήτων που θα ακολουθείται από μια αύξηση των κονδυλίων και τούμπαλιν. Σε αυτό λοιπόν έχουμε συμφωνήσει όλοι. Πολλές είναι οι τροπολογίες για τα χρηματοδοτικά πρότυπα, πολύ εύστοχες και στο πλαίσιο βέβαια των ε, δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τη δομή των υπηρεσιών αυτών θα πρέπει να εξετάσουμε και πάλι, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό 100% από τους ε, λαμβάνοντας τους αποδέκτες των υπηρεσιών, αν πρέπει να ακολουθεί ένα διαφορετικό πρότυπο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να λύσουμε βέβαια στο πλαίσιο της απαλλαγής, αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο ε, πρέπει να μας απασχολήσει και πάντως έχει νόημα να κατατεθεί η σχετική τροπολογία. Εν όλο πιστεύω ότι λόγω αυτών των πολλών ιδεών που βλέπω να συμπίπτουν μεταξύ των πολιτικών ομάδων θα είναι δυνατόν να επεξεργαστούμε ένα ικανοποιητικό για όλους κείμενο. Έκανα εγώ μια πρώτη προσπάθεια με τις προτάσεις μου. Την απέστειλα στις ε, ε, ομάδες Υπάρχει πρόταση για πιο ενεργό ρόλο για τις υπηρεσίες. Ε, εδώ δεν θα συμφωνήσω όμως, γιατί νομίζω ότι οι, δομ, δεν είναι δεν μπορούμε να δημιουργούμε νέες δομές για να επαληθεύουμε την τήρηση του δικαίου πάντοτε. Πρέπει να είναι ε, αυτό δουλειά της Επιτροπής και βέβαια των λοιπόν θεσμικών οργάνων. Οι υπηρεσίες έχουν ε, λόγο να κάνουν την ε, διακίνηση των πληροφοριών, ανακοινώσεων, απαντήσεων, ερωτήσεων, ε, να καταθέτουν δηλαδή μια σειρά θέσεων και προτάσεων και όχι να παρεμβαίνουν νομοθετικά. Αυτό άλλωστε είναι και το πεδίο πάνω στο οποίο κινούνται τροπολογίες επί το πλήστον. Ευχαριστώ λοιπόν σε όλους τους για την πληθώρα τροπολογιών. Ελπίζω να καταλήξουμε σε μια καλή και λογική λύση. Και βέβαια μετά από αυτό πρέπει να φροντίσουμε αυτό το οποίο θα αποφασίσουμε εμείς μεταξύ μας να γίνει και δεκτό από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού η οποία έχει την ε, διαχείριση της όλης εκθέσεως για τις, για τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά από πλευράς μου ως εισηγητή, καλό τους σκιώδεις εισηγητές και βέβαια τους λοιπούς συναδέλφους εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, όλοι Λουβτβίξον. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ και ως συζητητή για την εξαιρετική συνεργασία. Θεωρώ ότι Αυτά μας οδηγούν στη σωστή κατεύθυνση. Αν αναφερόμαστε στην αξιολόγηση του ελεγκτικού συνεδρίου για όλες αυτές τις ε, αρχές και το κατά πόσον ε, έχουν ε, ασχοληθεί νομότυπα και έχουν ε, φερθεί ορθώς όσον αφορά τι υποχρεώσει τους, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να αμφισβητήσουμε ε, το όλο ζήτημα και μπορούμε κάλλιστα να δώσουμε την απαλλαγή. Αν δείτε το σχέδιο κειμένου του συντάκτη της νομοδότησης και τι ε, προτάσεις για τροπολογίες για την εντολή, προσπαθούμε να εξεύουμε μια κάποια μορφή ισορροπία. Αφενός Σίγουρα η κάθε αρχή δεν μπορεί να δράσει πέραν της εντολής της και αυτό είναι σημαντικό να το επισημάνουμε και επίσης θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα πρέπει να εκμεταλλεύονται πλήρως την εντολή τους. Επομένως, θα πρέπει να λαμβάνουν τους πόρους που απαιτούνται για να διεξάγουν τα καθήκοντά τους. Και σε μια ειδική έκθεση ε, της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων, το ελεγκτικό συνέδριο δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι για να μπορέσει να εκτελέσει την εντολή της ε, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Ε, και αυτό φυσικά δεν ισχύει μόνο για την Αρχή Τραπεζών, αλλά και για τις τρεις αυτές αρχές. Και οι τρεις δεν λαμβάνουν αρκετά κονδύλια. Και δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Επίσης διαπιστώσουμε ότι ότι εξετάστηκαν και θέματα που αφορούν τους καταναλωτές. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες ε, για τις αρχές αυτές ώστε να μπορούν να είναι πιο δραστηρία σε θέματα προστασίας καταναλωτών. Κάτι το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε εδώ. Προσβλέπω λοιπόν στην συνεχή επικοδομητική εργασία επί του ζητήματος και είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε σε λογικούς συμβιβασμούς γιατί είναι εύκολο να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και και Σιγητά, βεβαίως, για τη δουλειά την οποία κάνατε. Θα είμαι σύντομος. Ε, η διάρθρωση την οποία αναφέρατε, πρώτα απ' όλα όσον αφορά τις γενικές παρατηρήσεις για τις εποπτικές αρχές. Εμείς δίνουμε βάρος ε, πως ε, τονίζεται ότι δημιουργήθηκαν αυτές οι εποπτικές αρχές για να συντονίζουν τη δουλειά των εθνικών εποπτικών αρχών και τονίζεται ιδιαίτερα η αρχή της επικουρικότητας, οπότε η διατύπωση που προτείνεται στη συμβαστική λύση α έχει τροποποιηθεί κάπως και έχει φύγει από μια έτσι, ουσιαστική λειτουργία και πάει περισσότερο προς μια λειτουργία προς την προσανατολισμένη προς τον σκοπό των εποπτικών αρχών. Μετά περνάμε στο μέρος δεύτερο προτεραιότητες ε, και εσωτερική διάρθρωση και εκεί πέρα θέλουμε και εμείς να γίνεται η οικονομία και θα πρέπει ακριβώς να χρησιμοποιούνται τα μέσα εκείνα τα οποία ε, διατίθενται σε εθνικό επίπεδο. Είναι επίσης πάρα πολύ θετικό το ότι απαιτείται την έκθεση να επικεντρωθούμε να επικεντρωθούν αυτές οι αρχές στην έντολή τους και να μην επεκταθούν παραπέρα. Επίσης, είμαστε κάπως επιφυλακτικοί για τις διατυπώσεις που έχουν σχέση με την υποχρηματοδότηση ήδη από την πρώτη φάση, γιατί αυτό προδικάζει ήδη μία προσαρμογή του προϋπολογισμού οπότε θα είμαστε κάπως πιο ε, θα ήμασταν εμείς κάπως πιο επιφυλακτικοί στις ε, διατυπώσεις μας ή θα μπορούσε και να φύγει τελείως η πρώτη περίοδος της συμβιβαστικής Β. Τα μοντέλα χρηματοδότησης που αναφέρεται μετά στο τρίτο μέρος, πράγματι είναι σημαντικό το ότι αναφέρονται στην έκθεση, αλλά θεωρούμε πως δεν μπορούμε να έχουμε χρηματοδότηση από ξεχωριστή γραμμή του προπολογισμού από τον προπολογισμό της Ένωσης, αλλά θα πρέπει το κόστος να το υπομιστούν ε, αυτοί οι οποίοι εποφελούνται από αυτή την εποπτεία, τα αντικείμενα δηλαδή αυτής της ε, εποπτείας. Άρα είμαστε σαφώς κατά του να διατεθούν εδώ πέρα κονδύλια από τον προπολογισμό και ζητάμε η διατύπωση αυτή να γίνει διαζευκτική, να πούμε είτε η, η συμβαστική δέλτα είναι η δέλτα και να χρηματοδοτούνται όπως είπα από αυτούς οι οποίοι υποφελούνται από την υποπτία μετά. Και με την επόμενη συμβασική θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην διατύπωση. Δεν πρέπει να προσπαθούμε να αποδώσουμε στις εποπτικές αρχές κάποιο είδους νομολογία. Σας ευχαριστώ. Νίλ Στόρβαλτς για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Το έχουμε συζητήσει αρκετά το θέμα ήδη. Οπότε θα προσπαθήσω να μιλήσω γερμανικά για να μην ε, το να μακρηγορήσω. Λοιπόν, έκανα, όπως είπα, κάποιες ε, προτάσεις οι οποίες ελπίζω να είναι αρκετά φιλελεύθερες. και νομίζω πως θα βρούμε κάποιους συμβιβασμούς για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, για να μην ταλαιπωρώ άλλο τους διερμηνείς, θα σταματήσω εδώ την άσκηση των γερμανικών. Α, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λιούκε κάτι κατάλαβε από αυτά που έλεγα και άρα κάτι έκανα. Ωραία. Σας κατάλαβα. Σας κατάλαβα και εγώ, λέω προς. Με συγχωρείτε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ενθάρρυνα τον κύριο Τόρβαλς να συνεχίσει. Ωραία. Και εγώ μια χαρά σας κατάλαβα, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, για την Γκουε Κύριε κύριος Κάρθη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την προσπάθειά σας ως συντάκτης αυτών των απαλλαγών. Υπάρχουν μια σειρά από θετικά στοιχεία και για την ομάδα μας το ουσιαστικό ζήτημα της Τραπεζικής Ένωσης και των φορέων που έχουν συσταθεί και πώς λειτουργούν είναι πολύ απαραίτητο. Θεωρούμε μια συζήτη, ότι είναι μια συζήτηση η οποία θα πρέπει να γίνει. Και αυτό κατά την άποψή μας δεν αντιμετωπίζει και δεν υπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών, υπηρετεί τις ανάγκες ε, άλλων και όχι των πραγματικών μας οικονομιών θέλουμε να υπάρχει η μέγιστη δημοκρατική συνεισφορά και εξετάσουμε τις γνωμοδοτήσεις μεμονωμένα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα του πραγματικού δημοκρατικού ελλείμματος, το οποίο κατά την άποψή μας ε, θίγεται εδώ, ε, υποσκάπτεται όλη η αρχή της επικουρικότητας από τις αρχές αυτές και από το γεγονός ότι οι πολίτες στα κράτη μάλες ε, θεωρούν ότι δεν ε, ε, τους ανήκει αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Η έκθεση αυτή και οι συμβαστικές τροπολογίες σε γενικές γραμμές μας βρίσκουν σύμφωνος, τις χαιρετίζουμε. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι πως κατά την άποψή μας οπωσδήποτε ως κοινοβούλιο πρέπει να έχουμε και αποφασίσαμε μια κοινή εντολή για τις ε, τρεις αυτές υπηρεσίες. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί τώρα γιατί απλά ε, εκπληρώνουν την εντολή που τους ε, δώσαμε. Το ίδιο και το δικαίωμα έκδοσης κατευθυντήριων γραμμών. Είναι τμήμα του υφιστάμενου κανονισμού για τις τρεις αυτές υπηρεσίες και μάλιστα στην περίπτωση της ΕΙΟΠΑ δηλαδή τους ασκούμε κριτική γιατί εργάστηκαν, ε, γιατί δεν υπήρχε όμνιμπους, μόνο ε, τους ότι δεν εργάστηκαν, αλλά δεν υπήρχε νομική βάση και κανονισμός όμνιμπους 2, οπότε επί σειρά ετών πρακτικά δεν ε, είχε λεπτομερείς αρμοδιότητες με βάση την νομοθεσία η υπηρεσία αυτή. Δηλαδή αν ε, έκανα ε, αυτά τα οποία ε, ζητάει εδώ πέρα η έκθεση θα πήγαινα στη Φραγκφούρτη, θα κοιτούσα τους ουρανοξύστες αλλά τίποτα πιο ουσιαστικό. Τώρα, για τον συντονισμό των υπηρεσιών θα πρέπει να σκεφτούν το τι σημαίνει αυτό και ποια είναι τα δικαιώματα περισσότερου συντονισμού δεν σημαίνει ότι θα τους ε, πάρουν την μπουκιά από το στόμα, αλλά όπου υπάρχουν διασυνοριακά προβλήματα και μπορούν να οργανώσουν κάποιες ε, συναντήσεις, ε, κάποια συνεργασία, κάποια αναρμόνιση, αυτό εγώ το βρίσκω σωστό. Αν δεν μας αρέσει μπορούμε να το πούμε. Το έχουμε κάνει και πρέπει να διατηρήσουμε το δικαίωμα Δυσάρεστη είναι η κατάσταση που είχαμε ζήσει όταν παραδείγματο χάρη κάποιο έχει την εντύπωση πως ε, προσπαθούν μέσω των ψηλών γραμμάτων να κάνουν διαρθρωτική πολιτική. Εκεί πέρα πρέπει να αντιδράσει το Κοινοβούλιο. Αλλά τώρα σε γενικές γραμμές αυτά τα οποία αναφέρονται δεν ξέρω θα είμαι πιο προσεκτικός. Γι' αυτό θεωρούμε πως ε, η ΕΕΠΑ 17 και η ΑΙΟΠΑ 11 μέχρι στιγμής καλύπτονται από τις ε, συμβασικές προτάσεις και οπωσδήποτε θεωρούμε πως οι υπηρεσίες αυτές ε, θα πρέπει να βρουν και προληπτικά στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή. Και δεν πρέπει να τις αποθαρρύνουμε με την έκθεση αυτή. Αλλά όπως είπα, γενικές γραμμές και τα λοιπά, εντάξει, μας βρίσκουν σύμφωνος. Και λέτε εδώ πέρα πως μπορούν να βγαίνουν και με λιγότερα λεφτά. Όποιος ε, τους ε, έχει επισκεφτεί ξέρει πως χρησιμοποιούν ελάχιστους πόρους και με αυτούς έχουν ε, εκδώσει πάρα πολλές κατευθυντήριες γραμμές. Και ενδιαφέρον θα ήταν να γνωρίζουμε τι θα κάναν δηλαδή με ακόμη λιγότερους πόρους. Ε, δεν ε, έχει επαφή με την πραγματικότητα αυτό. Η πραγματικότητα είναι πως οι υπηρεσίες αυτές έχουν ε, λάβει νομοθετική εντολή δεύτερου επίπεδου θα έλεγα και το αποτέλεσμα είναι τώρα πως έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις στο πλαίσιο, στην περίπτωση ΕΣΜΑ ας πούμε, που πλέον δεν μπορούν να εκπληρώσουν. Γιατί η ΕΣΜΑ πρέπει να κάνει κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει και τελικά θα βρεθούν να παρανομούν γιατί αντικειμενικά δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Και μετά το Κοινοβούλιο πρέπει να αποδίδει σωστά τις ευθύνε, Γιατί προσπαθούμε πάντα στους προπολογισμού να δώσουμε ε, περισσότερους πόρους. Τώρα, με λιγότερους ακόμα θα κάνουν ακόμη λιγότερο κομμάτι της ε, δουλειάς τους. Αυτό ισχύει οπωσδήποτε για την ΕΣΜΑ και για την ΕΙΜΑ μέχρι στιγμής. Και η ΕΟΠΑ θα δούμε τώρα. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλος να λάβει το λόγο, παρακαλώ. Ελίζα. Εγώ θα ήθελα απλώς ε, να επισημάνω κάποιες πτυχές οι οποίες ούτως ή άλλως αναβέρθηκαν και από τους αδέλφους που έλαβαν το λόγο πριν από μένα. Πιο συγκεκριμένα τα όσα είπε ο συνάδελφος ε, Λούντβικ και τα όσα είπε ο συνάδελφος ε, Σβεν Γίγκολτ. Οι αρχές αυτές, αυτοί οι οργανισμοί δεν ενδιαφέρονται να σταματήσουν, να υπάρχει συγκεκριμένο προπολογισμό, διότι ξέρουμε ότι ο προπολογισμό του προχωράει για χρόνια και ε, ξέρουμε ότι υπήρξαν αρκετέ ανεπάρκειε. Και όπω συμβαίνει πολύ συχνά και το αποδεικνύουν και οι αναλύσει μα άλλωστε. Πρέπει όμω να έχουμε κατά νου το εξή. Αυτέ οι αρχέ γεννήθηκαν πριν από μερικά χρόνια και πλέον βρίσκονται σε μια διαδικασία ε, σύστασή τους ε, και πρέπει ταυτόχρονα να αποδείξουν ότι έχουν υψηλή τεχνική ποιότητα ε, και να μπορούν να εφαρμόσουν πληθώρα νομοθεσίες η οποία δεν υπήρχε καθόλου στο παρελθόν. Εμείς λοιπόν στο μεταξύ έχουμε κάνει πάρα πολλά. Να υπενθυμίσω αυτό που έλεγε ο προηγούμενος πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και Νομισματικών Υποθέσεων. Προσπαθούσαμε να δούμε πόσα έγγραφα δημοσιεύτηκαν προσφάτως και είναι πάρα πολλά. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Επομένως, οι αρχές αυτές που είναι νέες αρχές και μόλις ε, συστήθηκαν και ίσως τη σύστησε και το κοινοβούλιο το ίδιο, τώρα λαμβάνουν εντολές, αιτήματα για πληροφορίες, για πράγματα τα οποία είναι ε, ζητήματα σοβαρής ευθύνης για να μπορέσουν να πληρώσουν τα κενά τα οποία ανοίχθηκαν στο παρελθόν. Το να λέμε λοιπόν ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τώρα τον προπολογισμό του ε, δεν ε, θα έχει κανένα αποτέλεσμα, διότι αν περιορίσουμε τον προπολογισμό αυτών των αρχών θα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες. Ουσιαστικά ε, θα υποσκάψουμε μόνοι μας αυτό που κάναμε, διότι θα μειώσουμε τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους αυτές οι αρχές. Αυτή ως πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά το στόχο της νομοθεσίας. Υπάρχει πλέον νομοθεσία. Πλέον όμως πρέπει να εφαρμοστεί και πρέπει να εφαρμοστεί με τον κατάλληλο τρόπο και πρέπει να υπάρχει αρμονία και συμβατότητα με την εσωτερική αγορά. Εμείς κάναμε πολύ μεγάλες προσπάθειες ε, προκειμένου να έχουμε μια οριζόντια νομοθεσία για αυτήν την εσωτερική αγορά. Ας δώσουμε λοιπόν τώρα τη δυνατότητα σε αυτές τις αρχές να δημιουργήσουν κατάλληλες προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους, να έχουν δηλαδή ένα κατάλληλο προπολογισμό. Και επίσης, οι άλλες πηγές εισοδήματος ε, ε, για τον προϋπολογισμό. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν περιορισμοί και για την εποπτεία αυτών των αρχών άλλωστε. Υπάρχουν περιορισμοί και για τη χρηματοδότηση αυτών των αρχών. Το κατανοώ αυτό. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε επιπλέον πόρους, μεν, αλλά θέλω να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί εάν ζητήσουμε από κάποιον οργανισμό, για παράδειγμα, να κάνει περισσότερες παρεμβάσεις. Και αυτό με λιγότερα χρήματα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και ε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας επί του θέματος αυτού, γι' αυτό και το ανέφερα. Ξέρω ότι δεν σας λέω και τίποτα καινούριο ή κάτι συγκεκριμένο, γιατί ούτως ή άλλως ακούστηκε ήδη και από τους συναδέλφους ε, στις προηγούμενες παρεμβάσεις αλλά βρισκόμαστε σχεδόν σε μια κατεπίγουσα κατάσταση και πρέπει να προστατεύσουμε το έργο αυτών των αρχών, διότι είναι νέες αρχές, τις οποίες ε, εμείς ε, θέσαμε σε αυτή την κατάσταση, Τους ζητούμε αποτελέσματα και πρέπει να βρουν έναν τρόπο να μας τα δώσουν αυτά τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ, δεν βλέπω να έχει στήσει κανείς άλλο στο λόγο. Ούτε είναι κανείς εδώ από τις υπηρεσίες. Καλά, τότε αλλάζω καπέλο γίνομαι εισηγητή, ε, συντάξει Σα ευχαριστώ θερμά για τι πολυάριθμε τοποθετήσει. Θέλω εδώ να υπενθυμίσω ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία τη απαλλαγή και όχι σε μια νέα διατύπωση τη νομική βάση των τριών υπηρεσιών, ούτε αναδιατύπωση μια βάσεω ε, χρηματοδότηση. Άρα, κοιτάω να καλύψω τα προβλήματα τα οποία μάλλον να αναφέρω τα προβλήματα τα οποία πρέπει μακροπρόθεσμα να επιληθούν, χωρίς όμως να προτείνω λύσεις για πράγματα που δεν μπορούν να λυθούν από αυτήν εδώ τη θέση. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση η οποία ναι μεν της καθιστά, ε, της ε, υπάγει στην τις, τις θέτει ανεξάρτητες ως προς τη λειτουργία τους, αλλά τις καλεί να βρουν και τρόπο χρηματοδότησης μόνες τους ε, οι υπηρεσίες αυτές. Βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να βρουν μια αγορά και εντός εισαγωγικών πελάτες για να χρηματοδοτηθούν. Αυτά ως ε, παρατήρηση παρεπίπτουσα. Μόνο μέσα από την, από την ε, αναθεώρηση του βασικού κανονισμού εσάς μπορεί να γίνει ε, κάποια αλλαγή και να λυθεί το ζήτημα, όχι μέσα από τις απαλλαγές. Αυτά λοιπόν νομίζω ότι μόνο με μια δημοκρατική ψηφοφορία μπορούμε να λύσουμε το ε, ερώτημα του μέχρι ποιο βαθμό μπορούν να φτάνουν οι κατευθυντήριες γραμμές Εγώ πήγα στο καινούριο κτίριο του Ιωβα στην ε, Φραγκφούρτη, το θαύμασα, φαινόταν πολύ εντυπωσιακό. Σε σχέση βέβαια με την ε, κεντρική τράπεζα που έχει πολύ πιο υψηλό κτίριο, δίνεται και η εντύπωση ότι μπορεί ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας να κοιτάει προς τα κάτω στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν είναι αυτό το ζητούμενο τώρα το θέμα αν θα μπορέσουμε να έχουμε ε, τις συμπράξεις που θα μπορούν να παρακολουθούν την λειτουργία και νομίζω ότι στο πλαίσιο μιας απαλλαγής το ζήτημα αυτό μπορούμε να το θέσουμε και πρέπει να τεθεί εάν μέσα από τις καθημερινές γραμμές προβλέπονται ζητήματα που δεν καλύπτει η νομοθεσία. Δεν λέω για τον κύριο Λάγκεν τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε τέτοιε περιπτώσεις. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ε, να αρχίζει να ορίζει προϋποθέσεις πράγματα στα οποία ακόμα δεν πραγματεύεται προσπαθώ να τα λέω στο δυνατόν πιο αφηρημένα. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε κάπου παρεμπιπτόντως και για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών επίσης. Έχει στην ε, στο σελίδα της ε, κάποιες οδηγίες, όχι κατευθυντήρες γραμμές, για τις εθνικές αποπτικές αρχές οι οποίες μπορεί να φαίνονται αθώες, οθόες, πολύ διακριτικές πάνω στη σελίδα. Για να το πω απλά, αλλά τελικά αποτελούν ιονή δεσμευτική, υποχρεωτική ε, οδηγία. Άρα τίθεται το ερώτημα σε ποιο βαθμό μπορούν να εκδίδουν και τις γραμμές και σε ποιο βαθμό μπορεί μια λογική της αυτορύθμισης να παραμένει ορθολογική εκδίδοντας οδηγίες και δευτερές γραμμές. Αυτό το έχουμε δει και με την PFIT 2 και με την ε, ε, EMIS, ε, με τις διάφορες οδηγίες για την πρόσκοπτη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών Υπάρχουν πολλές νομικές βάσεις, επαρκείς νομικές βάσεις για την ανάληψη εποπτικής ε, δράσης και για την ΕΠΑ, για τη τραπεζική ε, αρχή. Έχουμε την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ως επόπτη του επόπτη. Έτσι ορίζεται η ΕΜΠΑ, η Ευρωπαϊκή ε, Τραπεζική Αρχή. στο πλαίσιο τη της Ευρωζώνης παρακολουθεί εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, δρά με τρόπο ορθολογικό σε σχέση με τις ε, όσες τράπεζες έχει αναλάβει να εποπτεύει. Είναι τεράστιο το ζήτημα. Δεν είναι αμεληταίο και δεν μπορούμε, τουλάχιστον εγώ έτσι πιστεύω, να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι καταλήγουμε σε έναν μη υγιή ανταγωνισμό μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το ποιος έχει το πάνω χέρι και ποιος ορίζει τους ε, κανόνες. Πρέπει να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο λοιπόν για την δράση των ε, αρχών αυτών και αυτό δεν γίνεται με οδηγίες και εντολές. Εάν δεν ε, προχωρούμε παραπέρα από μια απλή διαπίστωση στη γνωμοδότηση αυτή είναι γιατί ξέρουμε ότι κάπου αλλού θα πρέπει να ρυθμιστεί. Απλώς ήθελα να το επισημάνω. Όπως είπα, ετοιμάζω, έχω αποστείλει μάλλον στους συναδέλφους των διαφόρων ε, ομάδων ε, συμβαστικές προτάσεις για τροπολογίες. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία επαφές. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε ταχύτατα να καταλήξουμε συνενετικά γιατί ξέρετε, σε σχέση με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού θα είμαστε ε, αποτελεσματικοί μόνο όσο είμαστε και ενωμένοι. Πρόκειται για το πρώτο δε κείμενο το οποίο έχουμε να διατυπώσουμε σε σχέση με τις υπηρεσίες και είναι σημαντικό να προχωρήσουμε με επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τη συζήτηση. Ψηφοφορία 23-24 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή. Ο έλεγχος του προπολογισμού προβλέπεται να ε, ψηφίσει στις 24 Φεβρουαρίου και λόγω των προθεσμιών που ορίζονται από τη συνθήκη η Ολομέλεια πρέπει να ψηφίσει την ε, ε, έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού στη δεύτερη Σύνοδο του Απριλίου. Αναλόγως βέβαια και οι τροπολογίες, έτσι ολοκληρώνει το θέμα αυτό. Τη ημερήσιας διάταξη. Κοιτάω να δω αν ο προσκεκλημένος μας βρίσκεται εδώ. Τον είχαμε προβλέψει για τις 5 στο σημείο 16 της ημερήσιας διάταξης. Έκθεση για το διάλογο σχετικά με την ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ Εάν δεν είναι εδώ λοιπόν ο προσκεκλημένο από την Επιτροπή, α κάνουμε μια μικρή διακοπή. Ένα λεπτάκι διάλειμμα για να μπουν οι εκπρόσωποι της Επιτροπής. Thank you very much indeed. We... Σας ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στο επόμενο ζήτημα της ημερήσιας διάταξης. Ενημέρωση από τον κύριο Λιβιέ Γκαρσόν, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Αρμόδιας Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα κάνει μια ενημέρωση για τα μέλη της Επιτροπής ε, ΕΚΟΝ για ε, τον τελευταίο διάλογο ε, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης που έγινε στη Ουάσιγκτον στις 13 Ιανουαρίου και περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία για τη συζήτηση και τη στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών για την εφαρμογή αυστηρών προτύπων κυρίως για το ε, χρηματοπιστωτικό ρυθμιστικό θεματολόγιο. Μετά από την παρουσίαση θα γίνει συζήτηση βάσει της διαδικασίας Catch the Eye. Να σας καλωσορίσω λοιπόν και να σας δώσω το λόγο. Ελπίζω να είναι σωστό το μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καθυστέρησα λίγο. Δεν έβρισκα και το δρόμο. Εδώ χάθηκα στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση λοιπόν, για να σας κάνουμε αυτή την ενημέρωση. Ε, είναι δύο φορές το χρόνο διεξάγεται αυτός ο διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Ο τελευταίος διάλογος έγινε πριν από μερικές εβδομίδες στις 12 Ιανουαρίου του 2015 στην Ουάσιγκτον. Ο τελευταίος είχε γίνει στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο. Και οι δύο αντιπροσωπείες έχουν δημοσιεύσει μια δήλωση, η οποία δημοσιεύτηκε στις 15 Ιανουαρίου, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, ε, ε, γνωστοποιήθηκε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν επικοδομητική η συνεδρίαση και έγινε σε θετικό κλίμα. Ήταν σαφές ε, ότι κυριάρχησε η συζήτηση για το καθεστώς ισοδυναμίας για τα παράγωγα τα οποία πηγαίνουν καλά, αλλά θα επανέλθω στο σημείο αυτό όταν ε, θα φτάσω στο κατάλληλο σημείο της ενημέρωσης. Είχαμε μια πολύ μεγάλη αντιπροσωπεία από όλες τις ε, βασικές αμερικανικές υπηρεσίες και πιο συγκεκριμένα από το ΣΕΚ, την SEC, την CFTC, FDIC, PPIOB και φυσικά τους συναδέλφους από το Υπουργείο Οικονομικών. να σας δώσω μία σύντομη αλλά πολύ συγκεκριμένη ενημέρωση και από εκεί και πέρα αν έχετε απορίες μπορώ να επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Το πιο ουσιαστικό τμήμα της συζήτησης ήταν το καθεστώς ισοδυναμίας των παραγόγων. Όπως γνωρίζετε, έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις με την Αμερικανική πλευρά εδώ και 1,5 χρόνο περίπου και οι συζητήσεις αυτές ε, είχαν σταματήσει με τον προηγούμενο πρόεδρο του CFTC, του ε, κύριο Γκένσλερ. Στη συνέχεια περάσαμε μια ενδιάμεση περίοδο ε, στην οποία έγιναν διάφορες προσπάθειες και υπήρξε κάποια πρόοδος ε, και ξεκινήσαν οι συζητήσεις με τον νέο πρόεδρο, το Tim Massent, τον Ιούλιο. Δεν έχουμε καταλήξει σε κάποιο σημείο στις συνομιλίες μας όπου θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις προκειμένου να θεωρήσουμε ότι υπάρχει ισοδυναμία. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ε, εγώ θα μεταβώ και πάλι στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα και κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν οι τελικές συζητήσεις. Η Αμερικανική πλευρά έχει προτείνει ένα σύστημα εξορθολογισμένης καταγραφής δεν μπορούν φυσικά να ε, μην έχουν καταγραφεί για τα ευρωπαϊκά παράγωγα στις ΗΠΑ γιατί αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει αμερικανικής νομοθεσίας αλλά έχουν προσφέρει μεγάλο φάσμα δυνατότητων ισοδυναμίας ε, βάσει των απαιτήσεων και τώρα συζητάμε τις λεπτομέρειες. Συζητούμε επίσης τις ε, ε, τη λειτουργία της επικουρικής αυτής συμμόρφωσης και αν υπάρχουν ερωτήσεις από πλευράς ΥΠΑ ε, αυτές να απευθύνονται στους επόπτες και όχι στους παίκτες της αγοράς απευθείας. Γι' αυτό ακριβώς βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Οι συζητήσεις ε, πηγαίνουν καλά, αλλά θεωρώ ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία επί του ζητήματος. Αυτή τη στιγμή έχουμε συμφωνήσει για τις παραμέτρους για το τι θεωρούμε ότι είναι ρυθμιστική διαφορά ε, η ΕΣΜΑ θα πρέπει να αναλάβει τα ενία για να κάνει κάποιες ε, πρώτες συζητήσεις για τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό οι βασικές αρχές ε, επί των οποίων να θεμελιωθεί αυτή η συνεργασία να αναφέρονται στην απόφαση για την ισοδυναμία. Αυτό ήταν ε, μακράν ε, το πιο σημαντικό ζήτημα στη συζήτηση. Η συζήτηση είναι ακόμα εν εξελίξη. Έχω κάνει κάποιες περαιτέρω τεχνικές ε, συναντήσεις απευθείας στη CFTC και κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν και περαιτέρω συζητήσεις την επόμενη εβδομάδα, διότι αυτή την εβδομάδα λάβαμε μια νέα υποβολή από την CFTC, η οποία είναι αρκετά ενθαρρυντική, αλλά πρέπει φυσικά να συζητηθεί διεξοδικά. Κατόπιν, κατά σειρά προτεραιότητας αν θέλετε ή ως προς το περιεχόμενο των συζητήσεων, το δεύτερο πιο σημαντικό τμήμα ήταν για τα benchmarks, όπου κατά βάση η ευρωπαϊκή πλευρά εξήγησε πού βρισκόμαστε στην νομοθετική διαδικασία με τους συνομοθέτες ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να προτείνει σχέδιο νομοθεσίας για τα benchmarks και φυσικά το ερώτημα που τίθεται είναι τι σκοπεύουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να εφαρμόσουν στη δική τους τη ε, ε, δικαιοδοσία τις αρχές της ΑΙΑΣΚΟ ε, δεν έχουν ακόμα διευκρινηθεί τα θέματα αυτά, επομένως ε, προσπαθούμε μέσω συνομολιών να δούμε κατά πόσον υπάρχει πρόθεση από πλευράς ε, Ηνωμένων Πολιτειών να ε, ψηφίσει νομοθεσία ώστε να μην υποχρεωθεί να χρειαστεί μόνο, να ανατρέχει μόνο σε ρύθμιση από τον ίδιο τον κλάδο όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Τρίτον, η εφαρμογή του κανόνα ΒΟΚΑ. Ε, η αμερικανική πλευρά μας ενημέρωσε και εμείς ε, τους ενημερώσαμε λίγο για το πού βρίσκονται οι συζητήσεις και στο Συμβούλιο και, στο, στο Συμβούλιο και στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αναδιάρθρωση των τραπεζών. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ελπίζουν να είναι έτοιμες και να είναι έτοιμες για την εφαρμογή μέχρι τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξετάζει και το κατά πόσον θα μπορούσαν να ε, υπάρξουν συνέπειες με την εφαρμογή του ε, νόμου Βόλκερ ε, και αν αυτό θα μπορούσε ίσως να δημιουργήσει προβλήματα. Όσον αφορά τους τίτλους, εξηγήσαμε γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει υψηλής ποιότητας ε, αγορά τίτλων ε, στην ευρωπαϊκή αγορά για να μπορέσουμε να έχουμε ε, διαφοροποίηση της οικονομίας κυρίως στις πλευρές, στις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ήταν δύσκολη χρηματοδότηση από τράπεζες και μόνον. Εξηγήσαμε ότι γίνεται μια απόπειρα να αναβιώσουμε την ανάπτυξη και φυσικά ζητήσαμε και υποστήριξη από πλευράς ΗΠΑ και διεθνών φόρα ε, για τα θέματα αυτά. Να σας πω ότι ήταν διαφορετική η αντίδραση από πλευράς ε, ε, του Federal Reserve και του Υπουργείου Οικονομικών. το Federal Reserve δεν ήθελε να υπάρχει καμία διεθνή δραστηριότητα στον τομέα αυτό γιατί θεωρούν ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις ΗΠΑ καταρχάς, επομένως δεν τους ενδιαφέρει και να προωθήσουν οποιοδήποτε διεθνές πλαίσιο για τους τίτλους, ιδιαίτερα αν θα είναι αυτοί αυτοί οι οποίοι θα πρέπει από εκεί και πέρα να σφραγίζουν τίτλους και να ε, δίνουν ε, κάποια ε, αξία σε υψηλής ποιότητας τίτλους αυτή ήταν ε, η δική του επιχειρομολογία. Ε, το ΔΕ Οικονομικών θεώρησε ότι μπορεί να είναι μεν ε, κατανοητό ότι μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το είδαν και από μακροοικονομική σκοπιά. Η αύξηση της ανάπτυξη τη Ευρώπης είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να βοηθήσει και να προωθήσει η Αμερικανική πλευρά. Σημειώσαμε την καλή συνεργασία στον τομέα των ασφαλιών Υπάρχει δέσμευση και από τις δύο μεριές για να ολοκληρώσουμε μια συμφωνία για να φύγουν ε, τα στοιχεία και να χρησιμοποιούνται σε εξασφάλιση της αντασφάλισεις. Ε, τώρα έχουμε ένα σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής από το Συμβούλιο. Η πλευρά των ΗΠΑ δεν χρειάζεται επίσημη εντολή αλλά πρέπει να ενημερώσουν οπωσδήποτε τον Ντότ Φρανκ και το νομοθετικό σώμα σε γενικές γραμμές υποθέτοντας πως θα λάβει η Κομισιόν κάποια διαπραγματευτική εντολή είπαμε πως θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις κάποια στιγμή τον Μάιο πιθανότατα επίσης σημειώθηκε καλή πρόοδος στον έλεγχο. Η σχέση μεταξύ των δικών μας υπηρεσιών και της PCAOB είναι πάρα πολύ καλές ε, και βελτιώνονται. Η Αμερικανική αντίστοιχη υπηρεσία συμφώνησε να παραπέμψουμε στην κοινή δέσμευση στην ε, δέσμευση που έχουμε να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο τους ελέγχους για να υπάρχει μια... να μπορούμε να βασιζόμαστε αμοιβαία ο ένας τον άλλον, κάτι το όταν επιτευχθεί θα είναι κάτι τόσο σοβαρό στην διεθνική συνεργασία. Πρέπει επίσης να πω πως ε, είχαμε την εμπειρία ε, για... Είχαμε την εμπειρία να μας εξηγήσουν το πόσο χαρούμενοι είναι που έχουν συμμορφωθεί με το πλαίσιο της Βασιλείας και το τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει ακόμα συμμορφωθεί. Βασικά τους εξηγήσαμε πως ε, ο κύριος όγκος ε, της διαφοράς μεταξύ των δύο δικαιοδοσιών αφορά το πώς αντιμετωπίζουμε τα CVA, κάτι το οποίο βεβαίω αυτή τη στιγμή είναι υπό εξέταση στην Βασιλεία, οπότε όταν ε, ολοκληρωθεί αυτή η εξέταση, οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμπεριλάβει τα αποτελέσματα αυτά στην ένομη τάξη της και άρα δεν θα υπάρχει πλέον αυτή η διαφορά και μετά για τα υπόλοιπα οι συνομοθέτες ε, είπαν πως θα πρέπει να αλλάξουν λίγο τις απαιτήσεις της ε, Βασιλείας και όπου συμβαίνει αυτό, αυτό γίνεται ε, για σοβαρούς λόγους και βεβαίως ε, σύμφωνα με την δικαιοδοσία που έχουν οι συνομοθέτες όπως θα έκαναν αντιστοίχως και είπα βεβαίως. Τέλος συζητήσαμε την ε, λύση μη τραπεζικών ιδρυμάτων, ε, το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη, και εκτός. Ε, όπως ξέρετε είναι και στο πρόγραμμα του Συμβουλίου Συστημικής Σταθερότητας. Είπαμε λοιπόν να καταλήξουμε σε μια κοινή πρόταση φέτος το συντομότερο δυνατόν. Το αφήσαμε ανοιχτό αυτό καθώς ακόμη συζητιέται στην ε, Κομισιόν και δεν έχει ακόμα ληφθεί κάποια απόφαση. Το εάν δηλαδή οι προτάσεις για την ε, λύση ή διάσωση άλλων μη τραπεζικών ιδρυμάτων θα γίνει ταυτόχρονα ή αργότερα. Τέλος, συζητήσαμε το ΤΙΛΑΚ η είπα μας ενημέρωσαν πως σκοπεύουν να το εφαρμόσουν πιθανότατα κατά τρόπο ισοδύναμο και ακόμη περισσότερο και βεβαίως μας ρώτησαν για τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς τους είπαμε πως ε, όσο μας αφορά η δική μας κατάσταση είναι κάπως διαφορετική γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα διαφορετικό πλαίσιο ονόματι MRL το οποίο θεωρούμε πως επαρκεί και βεβαίω θα θέλαμε το TILAC να αλλάξει ελαφρώς για να είναι κάπως πιο συμβατό με το MRL όχι λιγότερο αυστηρό, απλά πιο συμβατό έτσι ώστε να μην ε, υφίστανται οι τράπεζες ε, το να έχουν να προσαρμοστούν σε δύο ειδών προδιαγραφές και θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το Συμβούλιο Συντημικής Σταθερότητας μετά το ε, DIS για να το φέρουμε και στο Κοινοβούλιο και να πάνε και στο CIR για να εφαρμοστεί η TILAC. και εκεί πέρα ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις. Αν έχετε καμία άλλη ερώτηση είμαι στην διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω τον λόγο στους συναδέλφους, στον κύριο Λαμασούρ πρώτα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Διευθυντά, αγαπητέ φίλε, για την πολύ συγκεκριμένη και ενδελεχή αυτή έκθεση. Έχω κάποιες γενικές ερωτήσεις, καταρχάς κομισιόν. Ο κύριος με την προηγούμενη ο Μισελ Μπαγνή. μαζί με τον οποίο συνεργαστήκατε σε ρόλο κλειδί. Είχε ορίσει ένα φύλλο πορείας που κατέγραφε το σύνολο των κειμένων των οποίων είχε αναλάβει την πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσδιορίζοντας με τακτική μάλιστα επικαιροποίηση τη διαδικασία υιοθέτηση από την νομιθωτική αρχή των κειμένων που απέρεαν από τις αποφάσεις διαδοχικών G20 μετά την κρίση των Lehman Brothers. Από αμερικανικής πλευράς, κύριο κείμενο ήταν η Dot Frank, ο νόμος Dot Frank ένα κείμενο μακροσκελές, περίπλοκο, ασαφές, αδιαφανές, τουλάχιστον από αυτή την πλευρά του Ατλαντικού, από τη δική μας όχθη δηλαδή του Ατλαντικού, ήταν πολύ δυσνόητο, εκτός από κάποιους ειδικού λίγοι το καταλάβαιναν. Και η ερώτηση μου είναι η εξής. Έχουμε, έχουν περάσει κάποια χρόνια. Μπορούμε τώρα να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα για το τι έχει συμβεί στις ΗΠΑ από το νόμο Dodd Frank μέχρι τώρα. Γιατί στην αρχή τα πάντα φαινόταν να εξαρτώνται από τι συνθήκε εφαρμογή, τα εφαρμοστικά κείμενα και τον τρόπο με τον οποίο οι εποπτικέ αρχέ, που θα έπρεπε κιόλα να υποστούν τη δικασία τη μεταρρύθμιση, θα εφάρμοζαν στη συνέχεια τον νόμο Ντότ Φρανκ. Έχουμε λοιπόν μία ιδέα για την κατάσταση στι ΗΠΑ. Το νομικό πλέγμα δηλαδή που ισχύει. Μπορούμε να, να θεωρούμε ότι κάνανε το δικό τους μερίδιο των καθηκόντων που είχαν ήδη στη τελευταία ανάλυση ορίσει και που συνιστούσαν και στους G20 και στις θέσεις, τα κείμενα που έχουμε υιοθετήσει. Εμείς και εκείνοι από την πλευρά τους. Διαπιστώνεται περισσότερη σύγκληση ή μάλλον απόκληση. Και υπάρχουν αποκλήσεις οι οποίες μας δημιουργούν ε, αμηχανία αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φερέιρα ως συντονίστρια. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για την παρουσίαση. Μου φαίνεται πολύ σημαντική Και θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Ευθυντή να μας πει δύο λόγια παραπάνω, να μας δώσει πιο πολλές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθησαν αυτές οι διμερείς συνομιλίες. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει κινητικότητα, αλλά παραμένουν ακόμη αποκλήσεις και κενά σε σχέση με τις χρηματοπιστωτικές αγορές τις δύο του Ατλαντικού. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματεύεται τα θέματα αυτά, πώς τα επεξεργάζεται στο πλέγμα της TTIP. Γιατί έχει μια σειρά από στοιχεία, πολύ περίπλοκα όμως, στο πλαίσιο μιας γενικότερης συμφωνίας που φαίνεται να ε, διαγράφεται στον ορίζοντα ο χρηματοπιστωτικός τομέας τι θέση θα έχει. Θα είναι ένας ε, τομέας μεταξύ άλλων. Μεταξύ της ενέργειας, της έρευνας και ανάπτυξης, της γεωργίας και ούτω καθεξής. Ε, αν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Σε ποιο βαθμό εξασφαλίζει περιθώριο, ευελιξία και πώς ορίζει το σχετισμό μεταξύ αυτών των εργασιών και της TTIP. Γιατί προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι η στρατηγική μας ως Ευρώπη στο πλαίσιο αυτό. Αν θεωρούμε ότι πρόκειται για έναν τομέα ο οποίος πρέπει συνολικά να τύχει προστασίας, να ε, ε, ειδωθεί χωριστά από άλλες διαπραγματεύσεις ή αν θεωρούμε ότι θα πρέπει να στήσουμε κάποιες ε, περαιτέρω υποχωρήσεις από την άλλη πλευρά, ε, πρέπει να δούμε στο γενικότερο πλαίσιο τι ισχύει. Μπορείτε να μας ενημερώσετε. Καλά, ευχαριστώ κύριε Φανίφελ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν για την ενημέρωση. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση για τις συγκριτικές αξιολογήσεις γιατί προεξένησε έκπληξη αυτό το οποίο είπατε για προβλήματα με την ισοδυναμία και τις συζητήσεις με τρίτες χώρες. Για το ότι δεν υπήρχαν προθέσεις περί νομοθεσίες, στην ΕΠΑ και λέτε πως δεν έδωσαν σαφείς απαντήσεις. Ε, εγώ τους ρώτησα και μου ξεκαθάρισαν ε, πως δεν σκοπεύουν να έχουν προτάσεις ισοδύναμες με τη δική μας νομοθεσία. Μήπως να μας ενημερώσετε κάπως πιο λεπτομερώς για το τι συζητήσεις είχατε για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει το λόγο. Ναι, κύριε Ντεμπάκερ. Σύντομα να ευχαριστήσω και εγώ την Κομισιόν συζητάμε αυτή τη στιγμή νέα νομοθεσία για τις ε, συναλλαγές όσον αφορά την ε, χρηματοδότηση αξιογράφων, κάτι το οποίο βέβαια επηρεάζεται από τη χρήση εγγυήσεων. Το συζητήσατε αυτό επισήμως η ατύπωση με τους Αμερικανούς ομολογούς σας, ε, πώς το βλέπουν το θέμα. Ξέρω παραδείγματι σήμερα ότι κοιτάει το FSB σήμερα το τι γίνεται με λογιστικά πρότυπα για κουρέματα και άλλα τέτοια ζητήματα. Είναι κάτι το οποίο συζητάτε και στο δικό σας επίπεδο για να δούμε πώς θα υπάρξει κάποια τυποποίηση μεταξύ διαφόρων δικαιοδοσιών. Ευχαριστώ κύριο Σλάγγεν. Ευχαριστώ, δεν άφησα την εισαγωγή. Μια σύντομη ερώτηση μετά από αυτό το οποίο είπε η κυρία Φανίεν Χόιζεν. Τι γίνεται με την προσέγγιση με την έμια. Υπάρχουν κάποια ανοιχτά ζητήματα. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν ε, στο δεύτερο μισό της κυβέρνησης Ομπάμα τώρα που άλλαξαν τα πράγματα στο Κογκρέσο και την Γερουσία αν μπορούμε να υπολογίζουμε σε ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση να κάνω και εγώ μια ερώτηση για την συμπερίληψη των ε, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο TTIP. Θα ήθελα να γνωρίζω εάν ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής θα ήθελε να σχολιάσει για το πόσο πιθανό θεωρεί ότι θα είναι κάτι τέτοιο, να συμπεριληφθούν δηλαδή αυτές οι υπηρεσίες. Και στην περίπτωση που δεν συμπεριληφθούν, που ελπίζουμε να μην συμβεί, ίσως ε, να βρεθεί μια άλλη εναλλακτική λύση. Ευχαριστώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν. να απαντήσω στον κύριο Λαμασούρ, είναι σαφές ευθύς εξ αρχής ότι υπήρχαν ε, διεστάμενες απόψεις μεταξύ ημών και των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο το οποίο είχε ε, το πλεονέκτημα ότι μας έδινε μια συνολική εικόνα και από εκεί και πέρα να αρχίσουν να συμπληρώνουν. Εμείς ε, επιλέξαμε να πάμε κείμενο προς κείμενο τις συνομιλίες μας, ε, γιατί αυτό συνάδει περισσότερο με το νομικό μας πλαίσιο και τη νομική μας παράδοση και από ένα σημείο και πέρα ε, ήταν δύσκολο να βρούμε πού βρισκόμαστε γιατί ήταν τόσο διαφορετικές οι προσεγγίσεις που ήταν δύσκολο. Ε, όπως ξέρετε κύριε Λαμασούρ, εμείς έχουμε ε, καμιά εκατοστή εκτελεστικών πράξεων και πράξεων κατεξουσιοδότηση τις οποίες θα πρέπει να εγκρίνουμε και για κάποιες εξ αυτών Εάν δεν έχουν εγκριθεί, ε, στην πράξη η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται. Έχουμε λοιπόν ε, λίγο πολύ το ίδιο πρόβλημα με τους Αμερικανούς. Και αυτοί από πλευράς τους το έχουν λιγότερο από ότι εμείς, αν μου επιτρέπετε, διότι ε, εμάς η θεσμική μας δομή μας υποχρεώνει να έχουμε υψηλό βαθμό ε, εξειδίκευσης των ε, κανόνων στα κείμενα ε, πρωτογενούς και παραγωγού δικαίου, ενώ ε, πολλές φορές επειδή είναι πιο ομοσπονδιακό το σύστημα στις ΗΠΑ, εκχωρούν την εξουσία σε αυτούς οι οποίοι θα τα εφαρμόσουν. Εμείς ε, έχουμε μεν ε, κάποιο συντονισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών ε, και αυτών που εφαρμόζουν την νομοθεσία μας, αλλά πρέπει να δέωσουμε συγκεκριμένε οδηγίες για πολλά πράγματα, κάτι το οποίο έχει πλεονεκτήματα, αλλά έχει φυσικά και κάποια μειονεκτήματα και φυσικά αυτό επηρεάζει και το πόσο γρήγορα εργαζόμαστε. Αυτό που μπορούμε να πούμε, ε, είναι αρκετά περίπλοκο το ζήτημα, είναι ότι ε, για τα παράγωγα οι Αμερικανοί είναι πιο προηγμένοι, είναι ένα τομέα στον οποίο πυροχώρησαν πολύ πιο γρήγορα. Εμείς τους προλάβαμε όμως, κάτι το οποίο έρχεται και σε απάντηση του κυρίου Λάγκεν, που σχετίζεται και με μία άλλη ερώτηση που είχε τεθεί για το ίδιο ζήτημα. Στο τομέα των τραπεζών είναι το ίδιο. Ε, δεν είναι υποχρεωμένοι να περάσουν από νομοθετική διαδικασία. Ξεκίνησαν πιο αργά από εμά, γιατί δεν χρειάστηκε να γίνει όλη η συζήτηση που έγινε εδώ στα πλαίσια της ε, ε, ΣΕΑΕΡ και της σεαδ 4 και έφτασαν πολύ πιο γρήγορα στο ίδιο αποτέλεσμα με εμάς με μια ε, αρχιτεκτονική δομή εφαρμογής ε, των συμφωνών της Βασιλείας, ε, βάση των όσων περίπου είχαν γίνει και στη Βασιλεία, αλλά με διαφορετικά κείμενα, κάτι το οποίο εξηγείται φυσικά και σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο ε, εφαρμόζουν ε, τις ε, συμφωνίες αυτές από πλευράς ΗΠΑ. Ο καθένας βέβαια έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Αρκετές τράπεζες στις ΗΠΑ τις εφαρμόζουν αυτές, ενώ εμείς πρέπει να κάνουμε κάποιες προσαρμογές για τα τραπεζικά μας συστήματα, οι συνεταιρευτικές τράπεζες για παράδειγμα είναι μια τέτοια περίπτωση. Τώρα, ίσως το πιο ενδιαφέρον ζήτημα είναι το θέμα της ισοδυναμίας. Γιατί οι συζητήσεις που γίνονται για την ισοδυναμία σήμερα δεν απορρέουν από μια ε, διαφορετική προσδοκία. Όλοι προσπαθούμε να επιτύχουμε τον ίδιο στόχο. Και νομίζω ότι η σύσταση του G20 ήταν πολύ σαφής ε, στον τομέα αυτό και ε, η κάθε πλευρά το εφάρμοσε με πολύ εύστοχο και ειλικρινή τρόπο. Αλλά δεν συζητήσαμε επαρκώς ε, τα θέματα αυτά και επομένω η λογική τη εφαρμογή είναι διαφορετική και η προσέγγιση μα είναι διαφορετική. Εμεί έχουμε μια νομοθεσία, ενώ εκεί υπάρχουν δύο αρχέ, η CFTC και η SEC, οι οποίε εφαρμόζουν με πολύ μεγάλη διακριτική ευχέρεια τα κείμενα. Όπως γνωρίζετε, εδώ ε, η διακριτική ευχέρεια είναι πολύ δύσκολη, για να το πω έτσι, και δεν είναι και καθόλου επιθυμητή για την ε, νέα αγορά, ιδίως όσον αφορά τις εθνικές αρχές. Ε, επομένως ε, υπάρχει τελείως διαφορετικό επίπεδο. Ε, αντικειμενικά κατά πάσα πιθανότητα είναι πολύ ε, υψηλό σε ε, πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο, αλλά προσπαθούμε παρόλα αυτά να βρούμε μια λύση. Αυτό το οποίο εξαγωγό συμπέρασμα και νομίζω ότι με αυτό απαντάω και στην ερώτηση που ετέθηκε για το κατά πόσον συζητάμε ε, θέματα αυτής της μορφής είναι ότι θα ήταν προς το συμφέρον μας να βελτιώσουμε τη συνεννόησή μας για τα θέματα αυτά, ώστε να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί είμαστε στο στάδιο στο οποίο ε, εκπώνουμε κείμενα, αλλά καλό είναι πάντα να γνωρίζουμε ότι όσο πιο λογικά ε, ε, προσεγγίσουμε το ζήτημα και όσο πιο καλά προσεγγίσουμε τα θέματα, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσουμε να έχουμε ένα σύστημα ισοδυναμίας και θα μπορεί να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των επιποπτικών αρχών μας. Και είναι σημαντικό αυτό γιατί υπάρχει και η απόφαση των μη τραπεζικών ιδρυμάτων, κυρίως του CCP, διότι εκφύσεως αυτά είναι εξωτραπεζικά και μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με το CCP ε, και αυτό μπορεί να δημιουργηθεί και να οδηγηθεί στη συνέχεια σε συστημικό πρόβλημα και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα οι αμερικανικές και οι ευρωπαϊκές αρχές να ε, ε, προσπαθούν μέσω ψηφισμάτων να λύσουν τα προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται, θα πρέπει να δούμε ε, τι μπορούμε να κάνουμε για να διαγνώσουμε την κατάσταση και να έχουμε και κάποια μέσα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Με τις Αμερικανικές αρχές ε, αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε ε, πολύ νωρίς, ώστε να έχουμε και τις πρώτες ε, γραμμές ε, μιας νομοθεσίας, να δούμε αν έχουμε σύγκληση απόψεων, εάν διαβάζουμε με τον ίδιο τρόπο την κατάσταση, και να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε μια κοινή λογική και να υπάρχει μια κοινή διάγνωση της κατάστασης για να αποφύγουμε προβλήματα στο μέλλον. Αυτό φυσικά χωρίς να σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει το κείμενο το οποίο θα τους υποβάλουμε. Για τα benchmarks. Κατά πάσα πιθανότητα μας το έθεσαν όμορφα. Θεωρούν ότι η αυτορύθμιση είναι πολύ καλή και λειτουργεί αποτελεσματικά. Εμείς έχουμε διαφορετική άποψη. Θεωρούμε ότι η πρόσφατη ιστορία αποδεικνύει ότι δεν είναι και τόσο καλή και δεν λειτουργεί και τόσο αποτελεσματική και ότι πρέπει να υπάρχει ε, ένα αριθμιστικό πλαίσιο και να υπάρχει δημόσια παρέμβαση από αυτού. Ωστόσο, οι Αμερικανοί εταίροι μας δεν ε, είπαν σαφώς ότι έχουν οριστική θέση από αυτού. Δεν είπαν δηλαδή ότι ε, δεν θα νομοθετήσουμε τελεία και παύλα, ήταν λίγο πιο αμφίσιμη αν θέλετε. Και φυσικά εμείς τους επισημάναμε ότι εάν δεν υπάρχει νομοθεσία στις ΗΠΑ, τότε σίγουρα δεν υπάρχει βάση για μια διαδικασία ισοδυναμίας. Κάτι που θέτει και το ερώτημα για το κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχουν και ε, λύσεις εφεδρικές, ε, διότι μπορεί να είναι και προς το συμφέρον του ευρωπαϊκού κλάδου να μπορεί να βασιστεί σε ε, μη ευρωπαϊκά αμερικανικά benchmarks Δεν ήταν βέβαια στόχο αυτή τη συζήτηση να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα, τη συνεδρίαση, επομένω δεν τα συζητήσαμε. Για το ΕΜΙΡ ε, πήγα την επόμενη μέρα στο CFTC για να συζητήσουμε περαιτέρω τα ζητήματα. Δεν ε, έχουμε χρόνο συνήθω σε αυτέ τι συζητήσει και δεν είναι και το κατάλληλο βήμα για αυτέ τι συζητήσει, επομένω δεν συζητήθηκαν. Ο κύριος Λάγκεν χρειάστηκε να φύγει από ό,τι βλέπω. και νομίζω ότι είχα απαντήσει σε αυτό που ρώτησε στην αρχική μου παρέμβαση. Για να τα πω πιο λακωνικά, ο λόγος για τον οποίο ήταν πολύ περίπλοκες οι συζητήσεις και δύσκολες και επίπονες στο παρελθόν μεταξύ των δύο πλευρών ήταν συγκεκριμένο, αλλά φαίνεται ότι από τις αρχές του Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος μα έδωσε μια νέα όθωση από πλευράς Αμερικανικής και επομένω υπάρχει μια νέα διάθεση να καταλήξουμε σε μια μηδέα συμφωνία. Εμείς ε, κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να επιτύχουμε μια πρακτική λύση για τη διαδικασία καταχώρησης ε, και μας έχει μείνει το τελευταίο χιλιόμετρο. Ναι, μένει βέβαια είναι το τελευταίο, αλλά είναι και το πιο περίπλοκο και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και ελπίζουμε ότι στους επόμενους λίγους μήνες θα μπορέσουμε να έχουμε τα στοιχεία για να ληφθεί απόφαση ε, ισοδυναμίας σίγουρα πριν από την ε, ε, προθεσμία της 15ης Μαΐου. Και τώρα να περάσω στην ερώτηση της Ελίζα Φερέιρα. Η οποία σχετίζεται και με το δικό σας το ερώτημα κύριε Πρόεδρε για το TTIP. Το FMRD είναι καλό για την αμοιβαία πληροφόρηση, για να κατανοούμε καλύτερα ή για να ενημερωνόμαστε. Δεν είναι όμως ένα φόρουμ διαπραγμάτευσης για να επιλύουμε διαφορές δεν είχε αυτό το στόχο και βεβαίως όταν εκφράσετε τις ανησυχίες σας ερχόμαστε σε επαφή με τους Αμερικανούς ομολόγους μας αλλά δεν είναι αυτό το αντικείμενο υπό μία έννοια είναι ένα ήπιο μέσο γιατί μιλάμε πιο συχνά και χάνουμε έτσι σοβαρά αποτελέσματα. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να οδηγήσει ας πούμε σε ρυθμιστική σύγκληση μεταξύ Ένωσης και είπα... Υπ' αυτή την έννοια είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο είχαμε σκεφτεί στο πλαίσιο του TTIP και δεν θα το έλεγα εγώ δεύτερη λύση, γιατί είναι κάτι που έχει διαφορετική φύση. Χρήσιμο, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ειδικά όσον αφορά τη ρυθμιστική σύγκλουση σύγκληση, δεν δεσμεύει κανέναν. Πάρα πολύ συχνά, π.χ. όσον αφορά τα benchmarks, έχουμε μία θέση, έχουν αυτή άλλη θέση, δεν συμφωνούμε και τέλος. Εκεί πέρα τελειώνει το θέμα και έρχομαι άρα στο ερώτημα της κυρίας Φερέρα. Η θέση της Κομισιόν είναι σαφής ε, και θα είμαι εδώ πέρα πολύ προσεκτικός γιατί δεν είχαμε όπως ξέρετε εμείς την κύρια ευθύνη και οτιδήποτε γίνει στο πεδίο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών πρέπει να το δούμε στο παγκόσμιο πλαίσιο ε, των ε, διαπραγματεύσεων. Αλλά η θέση της Κομισιόν μέχρι στιγμής ήταν πως θα είναι επιθυμητό να ξεκινήσει μία συζήτηση για το κεφάλαιο αυτό της TTIP και θεωρούμε πως οι συζητήσεις αυτές θα πρέπει να έχουν ως στόχο και ρυθμιστική σύγκληση και πρόσβαση στην αγορά. Με άλλα λόγια δεν θεωρούμε ότι μπορούμε να συζητήσουμε πρόσβαση στην αγορά χωρίς ε, να συζητήσουμε τα ζητήματα ρυθμιστικής σύγκλησης. Για διάφορους λόγους, ένας εκ των οποίων προφανώς ε, βρίσκεται στην νομοθεσία που έχει περάσει το Κοινοβούλιο αυτό και αυτό σημαίνει πως ε, όλο το δευτερογενές αυτό δίκαιο σχετίζεται, συνδέει άμεσα το θέμα της ρυθμιστικής σύγκλησης με το θέμα της πρόσβασης στην αγορά. Γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε ισοδυναμία σε μια δικαιοδοσία τρίτου φορέα χωρίς να θεωρούμε πως υπάρχει ισοδύναμο με την δική μας νομοθεσία. Βεβαίως όταν μιλάμε για ισοδύναμο, μιλάμε για ισοδύναμο αποτέλεσμα. Δεν θα καλέμε εμείς τους άλλους τι θα κάνουν, αλλά τίθεται παρόλα αυτά ένα ζήτημα σύγκλησης των διατάξεων για να υπάρχει πρόσβαση στην αγορά για εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, Ε, για το TTIP και δεν γνωρίζω τώρα την στρατηγική που δεν έχει καν συζητήσει ακόμα το σώμα των επιτρόπων ούτε έχει δώσει κάποια κατεύθυνση αλλά ε, η θέση την οποία έχει εκφράσει η Κομισιόν είναι αυτή την οποία ανέπτυξα μετά. Μια άλλη ερώτηση ήταν το πόσο το πώς λαμβάνουν χώρα πρακτικά αυτές οι συνομιλίες ε, και πώς ερχόμαστε, πώς σχετίζονται με το TTIP. Δεν έχουν σχέση με το TTIP, συνεχίζονται όπως ε, γίνονταν πάντα, δηλαδή όποτε έχουμε ένα πρόβλημα αριθμιστικής σύγκλησης με τους Αμερικανούς συναδέλφους μας, προσπαθούμε να το λύσουμε προς το συμφέρον ε, των εταιριών, των δικών μας, και των δικών τους. Ε, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικοί κανόνες αλλά όχι δίπλοι κανόνες ε, και στο μέτρο του δυνατού προσπαθούμε να έχουμε μία όσο δυνατόν πιο ομαλή διατλαντική αγορά για τις ε, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προσπαθούμε να βασιζόμαστε ο ένας τον άλλον. Οπότε Όποτε υπάρχει ένα πρόβλημα, όπως με τα παράγωγα, όπως πιθανώς με τα benchmarks, ε, έχουμε άτυπες συνομιλίες για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Και η διαδικασία που κάνουμε π.χ. για τα παράγωγα δεν τον συνδέουμε, δεν το συνδέουν και οι Αμερικανοί με το TTIP ακόμα και αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία με το, για το TTIP για τις χρηματο ε, υπηρεσίες θα συνεχίσουμε εμείς γιατί όταν έχουμε βεβαίως επαφή δύο διαφορετικών σωμάτων θα έλεγα διατάξεων θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να λειτουργούν. Ποτέ δεν καταλήξαμε σε συνομιλίες σε κακή τυπίστη. Προσπαθήσαμε πάντα να λειτουργήσουμε στο μέτρο του δυνατού για να λειτουργούν οι αγορές με τρόπο που θα είναι ασφαλής χωρίς να τις επιβαρύνουμε ιδιαίτερα ταυτόχρονα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Τελειώσαμε με το σημείο 16 λοιπόν. 17. Διάφορα. Υποθέτω πως δεν υπάρχει τίποτα στα διάφορα. 18. Επόμενη συνεδρίαση. Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου από 3 το απόγευμα μέχρι 6.30 και την επομένη 9 με 12.30 και 3 με 6.30. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.